Uh, Αγαπητοί φίλοι, περιμένω τον κύριο Σιλικιώτη για να μπορέσουμε να αρχίσουμε με το σημείο 16 όπως είχαμε πει. Το αποφασίσαμε χθε αυτό, αλλά δεν είναι εδώ. Οπότε προτείνω να αρχίσουμε με το σημείο 14 στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για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 Πιστεύω, και φαίνεται αυτό και από τα στατιστικά δεδομένα, ότι αυτό το ζήτημα της ε, επανένταξης των εργαζομένων που αναρώνουν ε, σε ποιοτική απασχόληση αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Λέμε ότι συνταξιοδοτούνται οι άνθρωποι όλο και αργότερα στη ζωή τους, αλλά κατά πάσα πιθανότητα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της επαγγελματική του ζωής θα υποστούν κάποιο τραυματισμό. Η ιατρική βέβαια προδεύει. Άνθρωποι που είχαν κάποια σοβαρή ασθένεια ή κάποιο τραυματισμό τα ξεπερνούν αρκετά συχνά και έτσι έχουν τη δυνατότητα αυτής της επανένταξης χάρη στην ιατρική πρόοδο. Για μας λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τις χώρες μέλη είναι πολύ σημαντικό να επιτρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να επανεντάσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την περίοδο δηλαδή που βρίσκονται σε αποθεραπεία μετά από ένα τραυματισμό να φτάνουν στην επανένταξη στην επαγγελματική του ζωή. Όταν συνέτασα την έκθεσή μου προσπαθούσα βέβαια να σκεφτώ τι θα έπρεπε να συμπεριλάβω. Αυτά που υπάρχουν στο κείμενό μου σήμερα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να προχωρήσουμε παρατέρω. Είχα περιορισμένο βέβαια αριθμό λέξεων που μπορούσα να συμπεριλάβω, οπότε δεν τα έχω συμπεριλάβει όλα όσο θα ήθελα. Θα ήθελα λοιπόν με τροπολογίες να εμπλουτιστεί το κείμενό μου αυτό περισσότερο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει από μια σοβαρή ασθένεια ε, ή τραυματισμό μετά από ατύχημα για παράδειγμα τις περισσότερες φορές θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Θέλουν να βρουν τρόπο να επανέλθουν στην κανονικότητά τους. Σπάνια οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να επιστρέψουν. Πώς θα στηρίξουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα τους βοηθήσουν να επανενταχθούν. Θα το κάνουμε ή αντίθετα θα τους αφήσουμε να μείνουν σπίτι και να ακολουθούν μια εντελώς παθητική πορεία. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν ε, πολλές δυνατότητες να ε, επανεντάσσονται οι άνθρωποι αυτοί και πρέπει να το συζητάμε ανοιχτά και να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων. Και μια που μιλάμε για επιχειρήσεις, πρέπει να πω ευθύ εξ αρχής για τους εργοδότες ότι για αυτές τις βέλτιστες πρακτικές έχουμε την τάση να έχουμε στο μυαλό μας μεγάλες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει και ο δημόσιος τομέας. Δηλαδή, ακόμα και εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και αυτοί πρέπει να έχουν στήριξη και βοήθεια ώστε να μπορούν να επανενταχθούν στη δουλειά τους μετά από μια τέτοια μακρά απουσία. Χωρίζω την έκθεσή μου σε τρία τμήματα. Πρόληψη πρώτα απ' όλα. Σήμερα πολλοί εργοδότες σε πολλές χώρες επενδύουν στην πρόληψη. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό αυτό. Αλλά υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε έγκαιρες παρεμβάσεις, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε πιο αποτελεσματικά τον κόσμο. Τότε έχουμε και οικονομικά ωφέλη, γιατί όσο πιο νωρίς παρέμβουμε, τόσο πιο ήπιες είναι και οι συνέπειες μετά από ένα τραυματισμό. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με την ίδια την επανένταξη, την επιστροφή δηλαδή στον χώρο εργασίας. Όπως είπα, δεν μπορούσα να επεκταθώ πολύ λόγω περιορισμού του μεγέθους του κειμένου, οπότε αναφέρω εδώ μερικά μόνα μέτρα. Με στόχο να πω ότι ο κόσμος πρέπει να νιώθει ότι ο εργοδότης του το στηρίζει οι εργοδότες επίσης πρέπει να έχουν βοήθεια στη διάθεσή τους, ψυχολόγους και τα λοιπά, που να στηρίξουν τους ανθρώπους και μετά την απουσία αυτή να μπορέσουν να επιστρέψουν πράγματι στη δουλειά τους. Αυτά για την επιστροφή, όπου λέω επίσης ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει και ευελιξία για τον τρόπο που θα γίνει αυτό. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να αρχίσουν δουλεύοντας από το σπίτι. Επίσης θα μπορούσαμε εδώ να μιλήσουμε και για τις νέες δεξιότητες, γιατί αν κάποιος ε, βγήκε από τη δουλειά του και έλειψε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στην επιχείρησή του μπορεί να έχουν υπάρξει εξελίξεις στο μεταξύ. Άρα πρέπει να ενημερωθεί να αποκτήσει τις νέες δεξιότητες που χρειάζονται για να τα αποκριθεί στην νέα κατάσταση. Έτσι, σταδιακά θα μπορεί να αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζονται και να επανέλθει χωρίς πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το βάλουμε για τα, τις πρόσθετες δεξιότητες, νέες δεξιότητες και την κατάρτιση που ενδεχομένω χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Σε πολλά θέματα πρέπει να αλλάξουμε τη λογική μας. Δεν είναι βέβαια εύκολο, αλλά με εκστρατείες ενημέρωσης και συνειδητοποίησης αυτό μπορεί να γίνει. Και οι εργοδότες πρέπει να αντιληφθούν ότι και για αυτούς είναι προτιμότερο να επανεντάξουν τον εργαζόμενο που είναι έμπειρος, ακόμα και χρειαστεί να τον καταρτήσουν για λίγο, παρά να προσφύγουν σε κάποιον νέο που πρέπει να τα μάθει όλα από την αρχή, ένα νέο υπάλληλο. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε αποθεραπεία, είναι σημαντικό να μπορεί να έρθει σε επαφή με ειδικού, με ψυχολόγους, με γιατρούς εργασίας, οι οποίοι να είναι ειδικευμένοι σε τέτοιες περιπτώσεις και οι οποίοι θα ενθαρρύνουν τον άνθρωπο αυτό να επιστρέψει στη δουλειά του, εφόσον βέβαια η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει. Αυτή ήταν λοιπόν η εισαγωγή μου στην ε, έκθεση. Και συνοψίζω, όπως είπα και στην αρχή, και άλλα πράγματα θα ήθελα να προσθέσω στην έκθεσή μου και θα το κάνω με τροπολογίες. Ε, προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τους συναδέρφους, γιατί πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ επίκαιρη και πολύ σημαντική. Κανείς μας δεν ξέρει αν κάποια στιγμή βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή περάσουμε από κάποια σοβαρή ασθένεια ή τραυματισμό και αναγκαστούμε μετά από μια μεγάλη απουσία να επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παχ είναι σκιώδης ε, του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή της έκθεση που αποτελεί πολύ καλή βάση για τις περαιτέρω εργασίες μας. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε να κάνουμε με ε, πολλαπλά προβλήματα. Είναι επίκαιρο το θέμα και η έκθεση αυτή θα έχει μεγάλη αξία, κάτι με το οποίο συμφωνώ. Θα εργαστούμε πάνω στην εργασία αυτή προς όφελος ε, των πολιτών. Η εισηγήτρια αναφέρθηκε ε, στο θέμα του πληθυσμού και των αλλαγών ε, στην αγορά εργασίας. καθώς και κάποια φαινόμενα όπως είναι η ψηφιοποίηση που οδηγεί σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους μειοσκελετικές διαταραχές, ε, ψυχοκοινωνικές ε, πτυχές επίσης. Η συγγήτρια αναφέρθηκε στην πρόληψη που είναι και για μένα πολύ σημαντικό θέμα. Η πρόληψη ε, μπορεί να προλάβει ακριβώς τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Εάν κάποιος ε, ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχουμε συνεργασία από όλες τις πλευρές, εργαζομένους, ε, εργοδότες, ε, κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνική ασφάλιση κλπ. Δεν επιτρέπεται να αφήσουμε μόνο του έναν άνθρωπο που έχει βρεθεί σε αυτή την επισφαλή θέση. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε. Η εισηγήτρια Επίσης επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση και θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους ε, που λείπουν μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δουλειά τους ε, λόγω ασθενείας ή λόγω ασθενείας που σχετίζεται με την εργασία, αν και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει επικάλυψη των περιπτώσεων αυτών. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να υποστηρίξουμε την επιστροφή των ανθρώπων αυτών στον χώρο εργασίας και νομίζω ότι πολύ καλή προσέγγιση μπορεί να είναι αυτό που πρότεινε η εισηγήτρια, το να υπάρχει και ε, συνδρομία από διαφόρων ειδών υπηρεσίες Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αρκετά ε, άρρωστοι ώστε να πάρουν ε, άδεια αναπηρίας, από την άλλη δεν είναι σε θέση ε, να εργαστούν και να λειτουργήσουν σωστά στην αγορά εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι... Όπως είπε η συγγήτρια, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να εργαστούν, δεν θέλουν να πάρουν σύνταξη αναπηρίας. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να τους ξαναεπανεντάξουμε στην ε, αγορά εργασίας. Χρειάζεται να συλλέξουμε πολλές ε, πληροφορίες ε, και να εργαστούμε προς όφελος και των εργοδοτών και των εργαζομένων. Thank you. Then I'll give the floor Ευχαριστώ. Palmer από το S&D. Ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια έκανε εξαιρετική δουλειά. Μας παρουσίασε τα θέματα κλειδιά εδώ, καθώς και το πλαίσιο με το οποίο ασχολείται η έκθεση αυτή και ο σκιώδης συγητής αναφέρθηκε σε αυτό. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν στις δικές μου παρατηρήσεις θα επικεντρωθώ σε ε, σε τρία θέματα τα οποία θέλουμε να προσθέσουμε στην ε, έκθεση. Πολύ χαίρομαι που η συγγήτρια είπε ότι θέλει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η έκθεσή της ε, με τροπολογίες. Αυτό λοιπόν θα επιδιώξουμε να το κάνουμε σε συνεργασία μαζί της και τους άλλους σκιώδεις συγγητές. Εμένα το σημείο κίνησής μου στα θέματα αυτά είναι πάντα η αναγνώριση ότι ο καθένας από εμά, όλοι οι πολίτες σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαίωμα στην εργασία. Αυτό θεσπίζεται στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και στην ε, Οικουμενική Διακήρυξη ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους, να τους επιτρέψουμε να επανέλθουν στην ε, εργασία και να διατηρήσουν την εργασία τους. Αυτό είναι θέμα και δικαιωμάτων ε, και οικονομικό και είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη ώστε να φροντίσουμε να έχουμε τον κατάλληλο μηχανισμό για να στηρίξουμε τους εργαζομένους και άλλους εταίρους ώστε ο καθένα να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό άσχετα από την ηλικία του, άσχετα από το τι ασθένειε έχει, ε, τραυματισμούς ε, κλπ. Κάτι στο οποίο θα επικεντρωθώ στη δική μου δουλειά πάνω στην έκθεση αυτή είναι να φροντίσουμε ε, να υπολογίζουμε εξίσου την σωματική με την ψυχική υγεία, τη διανοητική υγεία, διότι ε, αυτό είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στον, ε, χρόνο, στον χώρο εργασίας. Ένας στους τέσσερις κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσει πρόβλημα διανοητικής υγείας, ψυχικής υγείας κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του. Βλέπουμε λοιπόν ε, νέες προκλήσεις στον τομέα αυτών. Βλέπουμε περισσότερους να παθαίνουν burnout, εξάντληση και κατάθλιψη. Και γι' αυτό Και Ακόμα και αν εργάζεται, ακόμα και αν δεν είναι κανείς στη δουλειά, νιώθει ότι είναι πάντα συνδεδεμένος με τη δουλειά λόγω του υπολογιστή του, λόγω των νέων μέσων. Με την έκθεση αυτή θα φροντίσουμε να προσέξουμε εξίσου ε, ε τις σωματικές ασθένειες και τραυματισμούς ε, με τα προβλήματα ψυχικής υγείας και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τελευταίο τμήμα της έκθεσης που μιλάει για αλλαγή της νοοτροπίας ε, διότι πρέπει να αλλάξουμε τη στάση της κοινωνίας και των ε, εργοδοτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, αντιμετωπίσουμε με θετικό τρόπο τα θέματα αυτά στο χώρο εργασίας. Ε, διότι έτσι θα συμβάλλουμε και στην καλύτερη αντιμετώπιση τους γενικά στην κοινωνία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε σε μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ατόμων με ασθένειες ε, και τραυματισμούς. Τους ε, ανθρώπους που έχουν χρόνια ασθένεια, διότι αυτοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη, ιδιαίτερες προκλήσεις. Κάποιοι από αυτούς επιλέγουν να εγκαταλείψουν ε, την εργασία τους, άλλοι όμως θέλουν να παραμείνουν ε, και για ε, οικονομικούς λόγους αλλά και λόγω της αξιοπρέπειας που συνδέεται με την εργασία. Ασχολούμαι αυτή τη στιγμή με μια καμπάνια που στόχο έχει να εισάγει νομική προστασία ώστε οι άνθρωποι με τέτοιες ε, ασθένειες ε, να ε, λάβουν συνδρομή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι άνθρωποι που έχουν καταληκτική μοιραία ασθένεια να μπορέσουν να παραμείνουν στο, χρόνο, στο χώρο εργασίας τους όσο θέλουν. Και το τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω αυτή τη στιγμή είναι η σημασία των εταιρικών σχέσεων ε, ώστε να βοηθάμε τους ανθρώπους να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας. Ε, σημαντικός φορέας εδώ είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ε, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ε, στο χώρο εργασία. Η έκθεση, όπω είναι διατυπωμένη αυτή τη στιγμή, δεν αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ε, θα προσπαθήσω λοιπόν ε, να το καλύψω αυτό σε τροπολογίε, διότι στα διάφορα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι μερικά από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα που επιτρέπουν στου ανθρώπου να επιστρέψουν στο χώρο εργασία μετά από ασθένεια ή τραυματισμό είναι τα προγράμματα όπου υπάρχει πραγματική συνεργασία ανάμεσα σε εκπροσώπους των εργοδοτών καταναλωτών και των εργαζομένων. Και ε, βλέπουμε πολλά παραδείγματα στα διάφορα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν να παίξουν ε, πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτών. Είναι ένας ρόλος τον οποίο έχουν παίξει με επιτυχία. Και αυτό ισχύει για τις ε, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Σημαντικό λοιπόν είναι να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην έκθεση. Κλείνοντας, ε, κύριε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και προσλέπω στη συνέχιση των εργασιών πάνω στην έκθεση αυτή, ώστε να υιοθετήσουμε μία έκθεση που να είναι όσο γίνεται φιλόδοξη για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επιστρέψουν στον χώρο εργασίας μετά από τραυματισμό ή ασθένεια και να αναγνωρίσουμε ότι αυτό δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό θέμα, είναι και θέμα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε μια πολιτική που να επιτρέπει στον καθένα να ε, απολάβει αυτού του δικαιώματος. Ευχαριστώ πολύ. Ο άλλος Σκιώδης δεν είναι εδώ και δεν έχει στείλει και αντικαταστάτη. Στην ΚΟΕ η Παλώμα Λόπες έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ ιδιαίτερο την εισηγήτρια για αυτή την ε, τόσο ε, σε σωστή στιγμή έκθεση. Θα ήθελα ε, να πω ότι συμφωνώ με την έγκαιρη πρόληψη και την πρόληψη ε, γενικότερα, γιατί αυτή είναι η σωστή γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Επίση, θεωρούμε ότι είναι σωστή η αναφορά που κάνει στα πλαίσια της ε, πρόληψη σε ένα εργαλείο πολύ σημαντικό, το οποίο έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η αναφορά στην υπηρεσία υγεία ή την όσα και ασφάλεια στην εργασία. Ε, ε, αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι συγκεκριμένα στοιχεία ε, όσον αφορά την επανένταξη και το σύστημα της επανένταξης. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει ιδιαίτερος να υπογραμμιστούν κάποια συγκεκριμένα θέματα και εκ των οποίων εγώ θα αναφέρω δύο. Πρώτα απ' όλα ε, θα πρέπει να δοθούν νέες δυνατότητες ε, και να βοηθήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες ε, τη στιγμή της επανένταξης. Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα αυτή η διαδικασία έχει εφεθεί στα χέρια κάποιων ταμείων ή κάποιων υπηρεσιών οι οποίες δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εάν ένας τραυματίας εργαζόμενος ε, προσπαθεί να ξαναενταχθεί ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ε, πρόσβαση σε ένα ειδικό σύστημα αδειών. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να το ίδιο το κράτος να το διαχειρίζεται. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα θέλαμε να θίξουμε Κοιτάξτε, εδώ δεν γίνεται συζήτηση για το τι μπορεί να βάλει κανεί μέσα σε μια έκθεση κτλ. Εν πάση περιπτώσει όμω καλό θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει μια αναφορά ε, σε εργαζόμενου που έχουν ε, αναπηρίε ε, και που επιστρέφουν μετά από άδεια, περνούν μια μεγάλη περίοδο ανεργίας ή αδράνειας. Εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμίσουμε ότι είναι θεμελιώδη σημασία να προσαρμοστούν και οι θέσεις εργασίας ε, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσει να επανενταχθεί ο εργαζόμενος ή εργαζόμενη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, έχουμε και πρακτικές ε, σωστές, έχουμε και καλά παραδείγματα, έχουμε συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες δημιουργούνται και στι οποίε προβλέπεται ιδιαίτερη υποστήριξη. Θα πρέπει οπωσδήποτε όμω να υπάρχουν και αρκετά κονδύλια έτσι ώστε να ε, υπάρχει η δυνατότητα ε, να παραμείνουν ενεργοί αυτοί ε, οι άνθρωποι οι οποίοι επανεντάσσονται. Και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο μας προβληματίζει η κατάσταση η οποία σχετίζεται με τη γύρανση του πληθυσμού. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πραγματική, την αντιμετωπίζουμε. Αλλά ε, ε, δεν είναι λύση η επιμήκυνση της εργασιακής ζωής των εργαζομένων. Υπάρχουν όντως εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να δουλέψουν. Για αυτούς λοιπόν θα πρέπει να ε, προστατευτούν τα δικαιώματά τους τη στιγμή που θέλουν εθελοντικά να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους και θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Δεν πρέπει όμως λόγω της γύρανσης του πληθυσμού να ε, προκύψει υποχρέωση επιμήκυσης της εργασιακής ζωής. Γιατί ε, διαπιστώνουμε ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Επιμηκύνεται η ζωή, η εργασιακή ζωή των πιο μεγάλων ανθρώπων ενώ από την άλλη μεριά έχουν μεγάλη δυσκολία και μεγάλα δυσκολία να μπουν στην αγορά εργασία οι νέοι και επομένως έχουν ε, μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Θα πρέπει να βρούμε στο θέμα αυτό την σωστή μέση λύση, δηλαδή να προσαρμόσουμε καλύτερα την ε, γενικότερη τοποθέτηση και γραμμή που ακολουθεί η έκθεση. Τέλος, πρέπει να ενισχυθεί η θέση ε, και ο ρόλος των, των κοινωνικών εταίρων, ιδιαίτερω δε των συνδικάτων. είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να ε, έχουν τη δυνατότητα τα συνδικάτα να έχουν λόγο σε όλες τις διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα, υγεία, ασφάλεια στους χώρους εργασίας κλπ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω να εκπροσωπείται εδώ η επόμενη ομάδα. Η πράσινη δεν είναι εδώ. Δεν εκπροσωπούνται. Η FDD, η Λάουρα Ατζέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ την συνάδελφο για την ε, πρόταση ε, γνωμοδότηση που μας κάνει. Εγώ συμμερίζομαι την γενική της τοποθέτηση. Ιδιαίτερος δε εκτιμώ το γεγονός ότι αφήνει πολύ περιθώριο μεγάλο περιθώριο έτσι ώστε ε, να έχει την δυνατότητα να εντάξει το αποτέλεσμα της κοινή εργασίας σε αυτό το έγγραφο που είναι τόσο σημαντικό. Ε, εξετίμησα ιδιαίτερο στο πρώτο ε, τμήμα και την σημασία και την υπογράμμιση που δίνεται στην πρόληψη έτσι ώστε να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να απευθυνθούμε στην καρδιά του προβλήματος που είναι ακριβώς ακριβώς ε, η έλλειψη πρόληψης ε, της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο και στη θέση εργασίας. Πολύ συχνά επαναλαμβάνουμε θέσεις ε, για αυτό το θέμα και είναι σημαντικό πλέον να το γράψουμε σε μια έκθεση. Είναι απαραίτητο ε, οι ε, επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν για την ασφάλεια στους χώρους και στις θέσεις εργασίας ε, και θα πρέπει να ακολουθήσουν και μία σειρά από στρατηγικά μέτρα για να αποφευχθούν οπωσδήποτε ατυχήματα αλλά και για να μην υπάρχουν πλέον εργασία, ασθένειες συνδεδεμένες με κακές και μη υγιεινές συνθήκες εργασίας. Το θέμα της έκθεσης σε καρκινογόνε ουσίες, ας πούμε, επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα εξισορροπιστικά και αποζημίωση, έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πραγματικά ε, σε τέτοιου είδους μέτρα από πλευρά των επιχειρήσεων. Ε, γιατί οτιδήποτε παθαίνουν, ας πούμε, οι εργαζόμενοι δεν αφορά στα πλαίσια πλαίσια της δραστηριότητάς μια επιχείρηση δεν, δεν αφορούν μονάχα τους ίδιους τους ε, εργαζόμενους αλλά έχουν μια σειρά ε, επιπτώσεων και σε ε, άλλους θα πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους ε, ε, εργαζόμενους που είτε παθαίνουν κάτι σε σχέση με τη θέση εργασία τους είτε έχουν ένα ατύχημα ή τους συμβαίνει ε, μια ατυχία. Εγώ είμαι Ιταλίδα, ξέρω πάρα πολύ καλά την πίεση που υφίστανται οι γυναίκες στην περίοδο της άδειας μητρότητας και πριν. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ασθένεια η μητρότητα ή η εγκυμοσύνη, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ατύχημα η εγκυμοσύνη και όμως ξέρουμε ότι τη στιγμή της εγκυμοσύνης, τη στιγμή της μητρότητας ε, οι γυναίκες ε, βρίσκονται αντιμέτωπες με την απόλυση, βρίσκονται αντιμέτωπες με προβλήματα, με πιέσεις, ε, πολύ συχνά μετατίθενται σε θέσεις λιγότερο σημαντικές από αυτές που κατήχαν πριν ή μετατίθενται σε άλλες ε, ακόμα και άλλες ε, πόλεις έτσι ώστε να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τη θέση εργασίας τους ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κάποια αναφορά στο θέμα αυτό. επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικό εντός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας να προβλεφθούν τα μέτρα αυτά τα οποία θα διευκολύνουν την επιστροφή στην εργασία και που θα διευκολύνουν βέβαια και την ίδια τη μητρότητα θα πρέπει να προβλεφθούν αναλόγως με το προφίλ του κάθε εργαζόμενου ε, και το προφίλ της επιχείρησης ε, κάποια, ε, κάποια προγράμματα κατάρτισης εκπαίδευσης και οπωσδήποτε και το είπε και η συγκήτρια πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούνται σε όλη τους τη διαδικασία και την διαδρομή τα άτομα αυτά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα έτσι ώστε το θετικός αντίκτυπος να είναι όχι μόνο ε, για τον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά το επαναλαμβάνω και για την ίδια την επιχείρηση πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, κινητροδοτήσουμε τους εργοδότες τις επιχειρήσεις να οδηγηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση και την διαδικασία και επίσης θα πρέπει να θέσουμε και τις βάσεις έτσι ώστε τα εργαλεία να είναι πολύ συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις ε, και κατά την έννοια αυτή και όχι μονάχα ε, για να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές ε, από χώρες που τις γνωρίζουν τις πρακτικές αυτές αλλά και για να έχουμε συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να ευνοήσουμε νέα εργαλεία εργασίας τα οποία θα είναι χρήσιμα όχι μόνο για να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές λόγω της μεταβιομηχανικής της εποχής μας, τις αλλαγές λέω στον εργασιακό ε, τομέα, ε, αλλά ε, για να μπορέσει να προστατευτεί και να παραχθούν χέγγια και για νέες μορφές εργασίας όπως είναι τα smart working κτλ και επίσης ε, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν την ε, δυνατότητα ε, να προσεγγίσουν τα εργαλεία αυτά ανάλογα με τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και τις δυνατότητες που έχουν. Θα πρέπει οι νέες μορφές, οι καινοτόμες μορφές εργασίας να καλυφθούν, να έχουν την απαραίτητη προστασία και κυδεμόνευση την οποία είχαν και οι παραδοσιακές μορφές εργασίας. Οποιαδήποτε κάλυψη ατυχημάτων ε, ή εργασιακών προβλημάτων θα διευκολύνει και τον κοινωνικό διάλογο. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε πίσω κανέναν. Κανένας δεν περισσεύει, κανένας δεν είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Ο καθένας εργαζόμενος και πολίτης είναι, αποτελεί σημείο ε, ε, πλούτου και επομένως θα πρέπει όλοι να προχωρήσουν μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και ε, να πω ότι εμείς δεσμευόμαστε να υποβάλουμε τροπολογίες έτσι ώστε ε, το τελικό αποτέλεσμα να είναι απολύτως αποτελεσματικό. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η υπόθεση αυτή για τις λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν ε, τους ε, εργαζόμενους μετά από μεκρά ασθένεια να επαναταχθούν στην εργασία τους έχει βέβαια νόημα. Η έκθεση ε, προσφέρει κάποιες βάσεις για εργασία και κάνει και κάποιες προτάσεις απόλυτα αποδεκτές με κάποιες μικρές εξαιρέσεις κατά τη γνώμη μας. Υπάρχει αυτή η βασική παρατήρηση όμως ότι δεν αφορά την Ευρώπη αυτή η υπόθεση αφορά τις χώρες μέλη και μόνο. Σε κάποια από τα σημεία σας αναφέρεστε στο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την εργασία μετά το 2020. Μα ειλικρινά όλα αυτά εξαρτώνται από τον κώδικα εργασία της κάθε χώρα μέλο. τον κώδικα εργασία, τον κώδικα κοινωνική ασφάλισης, των διατάξεων που ισχύουν μέσα στι επιχειρήσει και που τι έχουν συζητήσει με του κοινωνικού του εταίρου. Η Ευρώπη με τίποτα δεν πρέπει να προσθέσει ένα περιορισμό. Θέλω όμως να αναφερθώ στην ευθύνη της Ευρώπης για την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας. Μιλάμε για γενικά πράγματα όπως ακούσαμε και χτες για την διαφάνεια της εργασίας στην Ευρώπη και είδατε ποια είναι η αντίδραση των επιχειρήσεων που λένε φτάνει πια. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν και άλλους περιορισμούς, τεχνολογικούς, κανονιστικούς, φορολογικούς, άμεσους ή έμεσους με τα διάφορα μνημόνια που μας επιβάλλονται και τη λιτότητα. Έτσι κι αλλιώς θα παραμείνουμε σε έλλειμμα οικονομικά. Δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Και έπειτα υπάρχουν και κριτήρια που έχουν να κάνουν με του εργαζόμενου. Χθε είπαμε ότι οι γυναίκε πρέπει να δουλεύουν εφόσον θέλουν. Ναι, αλλά άμα δεν θέλουν, τουλάχιστον να μπορούν να μην δουλέψουν. Αλλά επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά μέσα σε δύο μέρε, ο μέσο όρο των μισθών και ο ελάχιστο μισθό που συγκλίνει προ την φτώχεια αναγκάζει τι γυναίκε να πάνε να δουλέψουν δημιουργώντας πολύ προβληματικές καταστάσεις στις οικογένειες. προκειμένου να αποκτήσουν κάποια αγοραστική δύναμη αποδεκτή. Όλα αυτά έχουν να κάνουν σε ένα μεγάλο βαθμό με τις διατάξεις της Ευρώπης. Η ανεργία δηλαδή δεν λέω ότι εξαρτάται μόνο από την Ευρώπη, αλλά φταίει η Ευρώπη σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν υπάρχει ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, σας θυμίζω. Κοιτάξτε τον κοινωνικό πίνακα του 2017. Αυξάνονται οι ανισότητες και ανάμεσα ε, τα δύο μέλη ενός ζευγαριού, αλλά και στις διάφορες χώρες μεταξύ χωρών, περιφερειών κτλ. Αν θέλουμε λοιπόν μια τέτοια βοήθεια πρέπει να τα έχουμε και αυτά υπόψη μας. Και έρχομαι και στους ηλικιωμένου. Υπάρχει ανεργία που βέβαια τους βαραίνει γιατί βλέπετε η παραγωγικότητα θέλει να μην κρατάμε ανθρώπους που κοστίζουν λίγο παραπάνω αλλά έχουν περισσότερη εμπειρία και από την άλλη μεριά πιέζουμε την ηλικία συνταξιοδότησης και τους κρατάμε στην αγορά εργασίας. Τελικά είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που αναγκάζονται να δουλέψουν για να πληρώσουν την ανεργία των εγγονών τους. Έτσι έχει φτιαχτεί το δικό μας κοινωνικό σύστημα. Συνεπώς, ναι, θα συνεργαστούμε και θα ε, προσπαθήσουμε να βάλουμε μια ισορροπία ανάμεσα στο κομμάτι που αφορά την Ευρώπη και αυτό που αφορά τις χώρες. Αλλά σας παρακαλώ για άλλη μια φορά μην μιλάτε εκ μέρους των επιχειρήσεων άμα δεν γνωρίζετε πραγματικά την κατάσταση που επικρατεί σε αυτές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, άλλος κανείς που θέλει το λόγο για αυτό το θέμα. Όχι. Ωραία, θα δώσω τότε το λόγο στην εισηγήτρια και πάλι. Παρακαλώ κύριε Ζιντάνσκα. Ή να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπω. Όχι. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους σκιώδες εισηγητές για τα σχόλιά τους. Όπως είπα και στην αρχή, είναι περιορισμένη η εκθεσή μου, το κείμενό μου. Περιορίζομαι από τους κανονισμούς. Γι' αυτό δεν έχω βάλει όλα όσα θα ήθελα να βάλω σε αυτή την έκθεση. Όμως να ξέρετε ότι θα ασχοληθώ σίγουρα με περισσότερα πράγματα μέσω τροπολογιών. Θα συμπεριλάβουμε και τους ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες που βρίσκονται σε τελικό στάδιο, για παράδειγμα, ε, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ κυρίως είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει από μια ασθένεια και θέλουν να επιστρέψουν στην εργασία τους. Αλλά θα το αναφέρω και αυτό. Θα κάνω μνήα γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Συμφωνώ. Επίσης, η έκθεση πρέπει να συμπεριλάβει τους κοινωνικούς εταίρους. Συμφωνώ και σε αυτό. Και αυτό ώστε η διαδικασία ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών να ισχύσει. Για τη Σλοβακία, για παράδειγμα, ε, τα συνδικάτα, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν την τάση να επικεντρώνονται περισσότερο στο διάλογο, στο θέμα των μισθών, περισσότερο παρά σε πράγματα όπως είναι αυτό που εξετάζουμε εδώ. Οπότε αν γνωρίζετε τέτοιε βέλτιστε πρακτικέ, ευχαρίστω να μου τι πείτε και να τι συμπεριλάβω. ξέρετε, α πούμε, ότι δικοί σα οι κοινωνικοί εταίροι ασχολούνται με αυτό το θέμα και προσπαθούν να βοηθήσουν ανθρώπου να επανενταχθούν στην εργασία του μετά από μια ασθένεια τραυματισμό, να μου το πείτε. Συμφωνώ επίση ότι όταν πρόκειται για μικρομεσαίε επιχειρήσει, πρέπει να διασφαλίσουμε οικονομική στήριξη απ' έξω. Γιατί δεν διαθέτουν ψυχολόγο, κότς ή ξέρω εγώ τι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε μπορεί να χρειάζεται όντως κάποιος εξωτερικός ειδικό να τις βοηθήσει. Και άρα πρέπει να βρεθούν οι πόροι. Και όχι μόνο. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι η στήριξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη. Δηλαδή δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε κονδύλια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει και οι χώρες μέλη να είναι σε θέση να στηρίξουν τέτοια βοήθεια από δικές τους οικονομικές πηγές. Κατά τα άλλα, είναι σημαντικό η βοήθεια να προσφέρεται. Αυτά που είπατε για νέες μορφές εργασίας επίσης θα τα συμπεριλάβω. Και πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο και με τα άτομα ε, με αναπηρίες γιατί βλέπετε ότι οι άνθρωποι που πέρασαν από μεγάλη διάρκεια απουσίας λόγω ή τραυματισμού μπορεί να επιστρέφουν με κάποια αναπηρία. Συμφωνώ. Σημαντικό όμως εδώ είναι να επικεντρωθούμε όχι μόνο στο άτομο που επιστρέφει, όχι δηλαδή μόνο στη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, αλλά και σε μια ρουτίνα που πρέπει να ακολουθεί η διαδικασία. Αυτό είναι σημαντικό για όλο το περιβάλλον που πρέπει να προσαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ τους σκιώδες και προσβλέπω σε συνεργασία μεταξύ μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Αυτή η υπόθεση όντως ε, απασχολεί πολλούς εδώ στην Επιτροπή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι, Κώστα Ντάβιτ, θέλετε να προσθέσετε κάτι μήπως, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, θα μπορούσα να πω λίγα λόγια. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, επικεντρώνεται στην πρόληψη. Οπότε αν, μπορεί να μην είμαστε στο άλλο άκρο, αλλά κοντά σε αυτό. Έχουμε κάποιες ε, ε, δραστηριότητες το, υπό την αιγίδα του Οργανισμού για την Υγεία και την ε, Ασφάλεια στην Εργασία EU OSHA. Πιστεύω ότι η έκθεση θίγει όλα τα σωστά σημεία. Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ε, εφαρμογή των βασικών αρχών. Ε, η έκθεση μιλάει για την οτροπία που επικρατεί και τις ε, και τις τοπικές παραδόσεις, διότι αν προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε την ίδια αρχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Πάντως η έκθεση αυτή εφιστά την προσοχή μας στην σοβαρότητα του προβλήματος. Οι εργαζόμενοι με προβλήματα υγείας ε, πρέπει να αναγνωρίζονται. Και νομίζω ότι τελικά αν δεν μπορούμε να εξετάσουμε τις, ε, την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, τουλάχιστον ε, να προσεγγίσουμε τον στόχο αυτό. Πάντως ε, εφιστούμε την προσοχή πολιτικών, ομάδων συμφερόντων κλπ. στο πρόβλημα αυτό το οποίο θα συναντήσουμε και στο μέλλον. Εγώ παρεπιπτόντως γιατρός είμαι. Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από τις ελλείψεις των πολιτικών υγείας. Ε, και άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι αυξάνεται συνεχώς το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων. Ε, με την τάση αυτή λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε επιδείνωση του προβλήματος. Κάποια κράτη-μέλη αυξάνουν συνεχώς ε, το όριο συνταξιοδότησης. Αναγνωρίζουμε πάντως τα πλεονεκτήματα της έκθεσής σας και θα προχωρήσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπα στην αρχή, έχουμε αναλάβει κάποιες δράσεις εμείς ήδη. Θα λάβουμε υπόψη μας τα συμπεράσματα του εγγράφου σας. και εμείς βρισκόμαστε υπό πίεση για να παρουσιάσουμε αποτελέσματα σε διάφορους τομείς. Ε, ελπίζουμε να τα δούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τις ε, παρεμβάσεις σας. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 25-26 Απριλίου και Κάποια στιγμή μετά από αυτό θα, θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια, δεν έχουμε όμως συγκεκριμένη ημερομηνία αυτή τη στιγμή. Θα ζητήσω από την Άγνες Ιονγκέριους ε, να προεδρεύσει, διότι ε, πρέπει να συναντηθώ με τον Υπουργό Εργασίας ε, της Αυστρίας. Η Αυστρία θα αναλάβει την προεδρία μετά την Βουλγαρία. Και θα συζητήσετε το σημείο 16 της ημερησίας διάταξης. Γιατί όχι το 15, δεν κατάλαβα. Ε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα γιατί δεν περνάμε τώρα στο σημείο 15 και λέτε ότι θα πάμε στο 16. Επαναλαμβάνω μιλητής, γιατί πάμε στο 16 και δεν κάνουμε πρώτα το 15 που είναι στη σειρά. κυρία Γιονγκέριος. Όπως ε, έχω καταλάβει, η πρόεδρος ήθελε το σημείο 16 να εξεταστεί στην αρχή της συνεδρίασης Άλλο ο δεν ήταν ακόμα εκεί, τώρα είναι. Και έχουμε 8 λεπτά πριν από το επόμενο σημείο. Αν συμφωνείτε λοιπόν θα κάνουμε τώρα το 16 και μετά θα κάνουμε το 15, οπότε θα είμαστε και στην ώρα μας. Εντάξει, λοιπόν, σημείο 16. Πρόκειται για τα εργασιακά δικαιώματα του πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού στην Κύπρο. ο εισηγητής πρώτα για να μας παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πρώτα πρώτα να απολογηθώ και να εξηγήσω στον συνάδελφο ότι είχα ζητήσει να συζητηθεί πρώτα το θέμα γιατί πρέπει να πάω στην Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας μετά. Ε, αλλά δεν ενημερώθηκε αν καιρά ότι θα έμπαινε πρώτον το θέμα για αυτή, αυτή η αλλαγή. Τώρα για το θέμα αυτό να πω ότι ενώ στην Ευρώπη Μιλούμε όλοι για την ανάγκη να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία. Ε, έθεσα αυτό το θέμα γιατί ε, στην Κύπρο υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την επισφάλεια του επαγγέλματο των ειδικών επιστημόνων. Αναφέρομαι στου διδακτορικού επιστήμονε διδασκαλία και έρευνα ε, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στι 30 Νοεμβρίου του 2017 καταθέσαμε γραπτή ερώτηση στην Κομισιό. Και το ερώτημα ήταν ότι ε, ε, θέσαμε ότι τα δικαιώματα ε, των διδακτορικών επιστημόνων διδασκαλία και έρευνα προστατεύονται από τη χάρτα του ερευνητή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το Euro Access, τα οποία φαίνεται να παραβιάζονται συστηματικά στο κρατικό πανεπιστήμιο τη Κύπρου, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στον τόπο. Η ερώτησή μα αναφερόντα τα βήματα που προτίθεται να κάνει η Κομισιό για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των διδακτορικών επιστημόνων και να αντιμετωπίσει ή να ζητήσει από την κυβέρνηση της Κύπρου να ρυθμίσει τις μη τυπικές μορφές εργασίας αυτού του είδους, ειδικά μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Πρέπει να πω ότι ενώ πέρασαν όλοι αυτοί οι μήνες δεν πήραμε καμία απάντηση από την Επιτροπή και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε χρήση του δικαιώματο να θέσουμε το θέμα στην Επιτροπή Απασχόληση του Κοινοβουλίου. Ε, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσία της εδώ και περιμένουμε την απάντησή της. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, παρά την αυξανόμενη ανάγκη για θέσει καθηγόντων, τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα στα Κυπριακά Πανεπιστήμια εκτελούνται συχνά από μη μόνιμους ερευνητέ, οι οποίοι ονομάζονται ειδικοί επιστήμονε. Απασχολούνται βάσει βραχυπρόθεσμο συμβάσιο... και σε πολλέ περιπτώσει η πληρωμή του καταβάλλεται με την ώρα. Ω αποτέλεσμα των ρομίσεων συμβάσεων εργασίας μερική απασχόληση και ορισμένου χρόνου, οι εργοδοτήμενοι δεν απολαμβάνουν κοινωνικά ωφελήματα, όπω άδεια ασθένεια, άδεια ανάπαυση, άδεια μητρότητα και πατρότητα. Δεν υπάρχει συνεισφορά του εργοδότη σε σχέδιο ιατροφαρμακευτική περίθευση. Κάτι που αποτελεί δυσμενή διάκριση σε σχέση με το υπόλοιπο ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και που ενδεχομένω αντίκειται και στην κείμενη νομοθεσία τη ίδια τη Κυπριακή Δημοκρατία. Επίση, λόγω έλλειψη εθνικού σχεδίου που να διέπει το επάγγελμα του ερευνητή, οι ειδικοί επιστήμονε δεν συμπεριλαμβάνονται επί του παρόντος των κατάλογων των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται από την αρμόδια ανεθνική αρχή. Και αναφέρομαι στο Υπουργείο Εργασία, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ω άλλο αποτέλεσμα, δεν υπάρχει σαφέ πλαίσιο για τον προσδιορισμό των ρόλων, των ευθυνών και των καθηκόντων των ερευνητών, καθώ και των εργοδοτών ή και των χορηγών του. Τέλο, οι ερευνητέ αυτοί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στι εκλογέ των πανεπιστημιακών χώρων και κάτι που αντίκειται στη χάρτα του ερευνητή. Ε, πρέπει να πω ότι ε, πολλοί από αυτούς του ερευνητέ ασχολούνται με ευρωπαϊκά ε, προγράμματα, προγράμματα δηλαδή που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συνδικάτο των ε, Διδακτικών Ερευνητών Διασκαλίας και Έρευνα ζητά την ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου του ερευνητή που να βασίζεται στην έδρα των ευρωπαϊκών προτύπων όπως η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή, ο Κώδικας Διοντολογίας για πρόσληψη των ερευνητών και οι κατευθυντήρες γραμμές του Access. Επιπλέον, το Συνδικάτο ζητά πλήρη πρόσβαση σε κοινωνικές παρχές όπως όλους τους εργαζόμενους. Άδειε ασθενείας και μητρότητας και άρση των περιορισμών όσον αφορά την επαναπρόληψη των ατόμων που εκτέλεσαν καθήκοντα διδασκαλία 30 μήνε σε διάρκεια 5 ετών. Πρέπει να πω πριν να ολοκληρώσουν του 30 μήνε, απολύονται από τα επαγγέλματά του. Γι' αυτόν τον λόγο πραγματοποίησαν και στι 22-23 του Ιανουαρίου 48 ε, ώρη απεργία. Εμεί θεωρούμε ότι αυτά τα αιτήματα είναι δίκαια. Περιμένουμε την τοποθέτηση τη ε, Επιτροπής ε, στο θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank Ευτυχώς είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσει να μας απαντήσει. Δίνω το λόγο στη Λούση Νταβονέ. Ζητώ συγγνώμη που δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις του συνάδελφου. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Νερ Πιάνσον από τη Γενική Διεύθυνση Ερευνών. Έρευνας. Και να απαντήσω καταρχάς όσον αφορά το θέμα που αφορά την έρευνα και η συνάδελφος θα ε, απαντήσει όσον αφορά την αγορά εργασίας. Καταρχάς, ε, είδα την ερώτηση, έχουμε απαντήσει. Βρίσκεται καθοδόν προς το Κοινοβούλιο η απάντηση. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι εδώ έχουμε δύο θέματα. Καταρχάς, την πολιτική της αγοράς εργασίας και τις προϋποθέσεις και κατόπιν ε, έχουμε τα συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τους ερευνητές. Εγώ λοιπόν μπορώ να απαντήσω σε αυτό που αφορά τους ερευνητές και τα πανεπιστήμια. Έχουμε λοιπόν μία σύσταση και πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για σύσταση, όχι για κανονισμό. Ε, από το 2005. Η σύσταση λέει να καθιερωθούν καλές συνθήκες εργασίας για τους ερευνητές, να έχουν τις ίδιες συνθήκες απασχόλησης με άλλους, να είναι διαφανείς οι συνθήκες απασχόλησής τους. λόγω των προσόντων τους και αυτή είναι μία σύσταση που έχουμε εκπονήσει. Από εκεί και πέρα εναπόκειται απολύτως στο Πανεπιστήμιο να αποφασίσει υπό τι προϋποθέσεις θα απασχολεί το προσωπικό του. Δεν μπορούμε λοιπόν να επέμβουμε σε αυτό. Είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες στοιχείες που αφορούν την αγορά εργασίας. Ε, θα απαντήσει η συνάδελφο σε αυτές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχο έχει να ε, ξεκινήσει μία πρωτοβουλία για τις ασφαλείς ε, συνθήκες απασχόλησης ε, που θα παρουσιαστεί κατά την επόμενη διαβούλευση του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Και η ανησυχία που οδήγησε στην πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό που συζητάμε εδώ, ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη που δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης, είτε μιλάμε για περιπτώσεις ασθένειας, για άδεια μητρότητας, για σύνταξη κλπ. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα χαρτογράφησης ε, που κάναμε το 2017. Επίσης είχαμε διαβούλευση σε δύο στάδια των κοινωνικών εταίρων πάνω στο θέμα αυτό και ξεκινήσαμε και μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση. Ω αποτέλεσμα τη διαβούλευση αυτή και τη χαρτογράφηση που κάναμε, σκοπεύουμε ε, στα μέσα Μαρτίου ε, να ξεκινήσουμε την πρωτοβουλία αυτή που θα εφαρμόζει την αρχή 12 του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που λέει άσχετα από το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης ε, για ε, υπαλλήλους ε, αλλά και αντιστοίχω και για τους αυτοαπασχολούμενους θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα πρόσβασης σε κοινωνική προστασία. Συνεχίζουμε τις έρευνές μας στο θέμα αυτό και με την πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να καλύψουν τα κενά που εντοπίσαμε όσον αφορά την κοινωνική προστασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτώ λοιπόν τον συνάδελφο που έθεσε την ερώτηση. Θέλετε να επανέλθετε ή σας ικανοποιεί η απάντηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να πω ότι η Επιτροπή μας ε, σε πάρα πολλέ εκθέσει τον προηγούμενο χρόνο ασχολήθηκε με τα θέματα τη επισφάλεια στην εργασία και των άτυπων μορφών εργασία ε, και είναι ένα θέμα που αναμένουμε βεβαίω ε, από την Επιτροπή. Χαιρετίζω για αυτήν την πρωτοβουλία που αναφέρεται για την εφαρμογή της αρχής 12 του Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τη σύσταση στα κράτη-μέλη να καλύψουν τα κοινά. Θα αναμέναμε όμως από την Επιτροπή ε, και στα θέματα της αγοράς εργασίας και στα θέματα ε, των ερευνητών ε, να γίνει σύσταση ε, και προς την κυβέρνηση της Κύπρου αλλά και προς το ίδιο το ε, δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο είναι κρατικό ε, το να εφαρμόζει αυτές τις συστάσεις δηλαδή αυτά που αναφέρθηκαν εδώ θα αναμέναμε ότι θα μπορούσε να γίνει με μια σύσταση και προς την κυβέρνηση και προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου ώστε να νιώθουν μια μεγαλύτερη πίεση για να εφαρμόσουν πραγματικά και το χάρτα, το των κοινωνικών δικαιωμάτων αλλά ε, και τις ε, συνθήκες απασχόλησης των ερευνητών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από ό,τι κατάλαβα, η γραπτή απάντηση βρίσκεται καθοδόν, κάπου ανάμεσα στο δικό σας στήριο και το δικό μας. Θα έχετε λοιπόν αργότερα την ευκαιρία να δείτε πώς ε, μπορείτε να συνεχίσετε πάνω στο θέμα αυτό. Τρία λεπτά καθυστέρηση έχουμε. Προχωράμε στο σημείο 5 της ε, κατευθυντήριες ε, γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Το σημείο 15. Είναι παρούσα η συγγήτρια. Κυρία Στανόκα. Να σας δώσω το λόγο, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελεί για μας ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπογραμμίζονται περισσότερο τα κοινωνικά δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες, η κοινωνική προστασία, η μείωση των αποκλεισμών και μιλάμε επίσης και για ελάχιστο μισθό. Είναι λοιπόν αυτό το οποίο το Κοινοβούλιο μας ζητά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και με ικανοποίηση διαπιστώσαμε στην πρόταση της Επιτροπής ότι περιλαμβάνεται και ο όρος ε, ε, απασχόληση ποιότητας και όχι απλώς απασχόληση όπως γινόταν μέχρι τώρα. Το σημαντικό λοιπόν είναι η σύνδεση με το κοινωνικό πυλώνα που περιλαμβάνεται στο εξάμεινο και στις ε, συστάσεις αναχώρα. Επίσης περιλαμβάνεται στο κείμενό μας πιο συγκεκριμένα η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφή ένδυας για να δημιουργήσουμε δικαιώματα για περισσότερο ακόμα κόσμο στην αγορά εργασίας, κοινωνική προστασία και να τονίσουμε περισσότερο την απασχόληση ποιότητας και την αγορά εργασίας για όλους. Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι υπηρεσίες κατάλληλης φροντίδας, προσβάσιμες και όχι ακριβές είναι κάτι που πρέπει να έχουμε. Είτε πρόκειται για τα παιδιά, είτε πρόκειται για εξαρτώμενα άτομα. Θα θέλαμε αυτό να υπογραμμιστεί περισσότερο στο κείμενο. Όμως πρέπει να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικά δημοκρατικός έλεγχος στη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί μόνο σε αυτό το θέμα, ενώ ζητάμε πλήρη συμμετοχή. Μα ζητούν τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμεί όμω θέλουμε να λαμβάνονται και υπόψη. Όχι όπως έγινε τις προηγούμενες χρονιές που τα βάλανε σε ένα σερτάρι. Υπάρχει δημοκρατική διαδικασία, διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, κάτι το οποίο είναι πολύ καλό βέβαια. Και τους ευχαριστούμε. Οπότε τώρα θα ήθελα να ακούσω τους κοιόδες εισηγητές, να μου πούνε τι πιστεύουν για την πρότασή μας. και θέλουμε τη στήριξη της Επιτροπής Απασχόλησης έτσι ώστε με δυνατή φωνή να προχωρήσουμε και να μας λάβουν υπόψη τους και στην Κομισιόν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Σάτμαν έχει το λόγο, από ό,τι κατάλαβα. Εσείς μιλάτε εκ μέρους του ΕΛΚ, σωστά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Γιατί θα πάρω εγώ το λόγο αντί και τον κύριο Πλούρα που δεν μπορούσε να είναι. Είναι σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών αυτή τη στιγμή για τα άτομα με αναπηρία και μου ζήτησε να διαβάσω την ε, θέση του. Οπότε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ την κυρία Σδανόκα για την ε, έκθεσή της. Ε, συμφωνούμε που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σίγουρα η τα κοινωνικά δικαιώματα, οι συζητήσεις με τους κοινού, κοινωνικούς εταίρους είναι μια πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε. Οι δικές μου τροπολογίες τώρα έχουν σαν στόχο να προσθέσουν κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, η στήριξη των μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, απλούστευση και απαλλαγή από το διοικητικό άχθος. Αυτό επίσης που είναι πολύ σημαντικό είναι να στηρίξουμε την ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε απαιτήσει για πλήρη απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες. Αυτή η ομάδα πολιτών, που είναι 80 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα, αποτελούν ένα τεράστιο δυναμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οικονομική ανάπτυξη και υπέρ της κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Οι χώρες μέλη επίσης και η Επιτροπή πρέπει να προωθήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για μια ανοιχτή αγορά εργασίας. Χρειάστηκε αναθεώρηση ε, των συστημάτων που αποφασίζουν προκειμένου ακριβώς να είναι ανοιχτή αγορά εργασίας. Τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να μπορούν να έχουν βοήθεια από συμβουλευτικές υπηρεσίες. Χρειάζεται επίση στήριξη και στους ανθρώπους που φροντίζουν τέτοια άτομα. Να μην έχουν ε, περιορισμό για τη δουλειά τους. Μόνο έτσι θα μπορούν και τα άτομα με αναπηρίες να συνεχίσουν στην αγορά εργασίας. Οι κατευθύνες γραμμές πρέπει να στηριχθούν επίσης από τα διευθυντικά ταμεία, δηλαδή και από το κοινωνικό ταμείο. Συνεπώς, αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Πλούρα που σας παρουσίασα μόλις τώρα. σας ευχαριστούμε κύριε Χάτμαν. Τώρα, να δώσω το λόγο στον κύριο Τέτσον από τους σοσιαλιστές. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το πολύ καλό σχέδιο έκθεσης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόληση. Το πρόβλημα είναι η ε, τροπολογία 4. Αυτή είναι καθοριστική σημασία για το σύνολο της έκθεσης. δεν ε, έχει γίνει η σωστή διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η τελευταία αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών έγινε αφού αγνοήθηκε τελείως ε, η γνώμη του Κοινοβουλίου και αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Θα πρέπει με δημοκρατικό τρόπο και με πλειοψηφικέ αποφάσεις ε, να διαμορφώνονται οι πολιτικές. Άλλωστε είναι και προ συμφέρον ε, και του Συμβουλίου να συμμετάσχει σωστά το Κοινοβούλιο. Διότι εάν και το Κοινοβούλιο συμμετέχει, αυξάνεται η νομιμότητα και η αποδοχή ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και τα δύο αυτά είναι εργαλεία για τον ευρωπαϊκό συντονισμό στον τομέα της ε, αγοράς εργασίας. Το σχέδιο έκθεσης ε, συμπεριλαμβάνει 25 τροπολογίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις μηδενικού χρόνου, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς το S&D. Και γι' αυτό το επικροτούμε. Θα θέλαμε πιο ισχυρή διατύπωση όσον αφορά ε, το ελάχιστο εισόδημα. Οι εργαζόμενοι αποτελούν τουλάχιστον, αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το μισό της οικονομίας. Τα κοινωνικά τους δικαιώματα λοιπόν θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να μιλάει με μία φωνή όσον αφορά το δικαίωμα συναπόφασης και γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω όλες τις πολιτικές ομάδες από κοινού να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και προτού να δώσω το λόγο στο ECR. Να σας πω ότι έχουμε μία ομάδα προσκεκλημένων στο πίσω μέρος της αίθουσας. Είναι προσκεκλημένοι του συναδέλφου Μάσιμο Παουλούτσιο και έρχονται από τον Δήμο του Αμπρούτσο. Σωστά είναι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Καλώς ήρθατε στην ομάδα μας. Ε, Ε, το ECR δεν θέλει να πάρει το λόγο ε, εκ μέρους του ECR. Όχι, τότε δίνω το λόγο ε, στην συνάδελφο Τουμ εκ μέρους της ομάδας ALDE. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Στάνοκα συνέταξε εξαιρετική έκθεση και απλά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιους συλλογισμού σχετικά με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, την κατευθυντήρια γραμμή 8 που έχει να κάνει με τις ίσες ευκαιρίε. Πιστεύω ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων είναι κλειδί ε, για να προωθήσουμε τις ίσες ευκαιρίες ε, και θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι διακρίσεις υπονομεύουν τη σωστή λειτουργία της αγοράς εργασίας και εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Οι διακρίσεις ε, λοιπόν ε, έχουν πολύ υψηλό τίμημα. Ε, δεν είναι όμως αποτελεσματικές ε, οι μέθοδοι για την καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδιαίτερα όχι σε επίπεδο κρατών μελών. Ε, σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου νομολογία που οφείλεται σε χαμηλή αποτελεσματικότητα των σχετικών φορέων. Οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής ή λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων ε, είναι ε, μεγάλο πρόβλημα και ιδιαίτερα μεταξύ μεταναστών και προσφύγων. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε διακρίσεις στην αγορά εργασίας και περιορίζεται και η ελευθερία κινητικότητας. Και οι διακρίσεις λόγω ηλικίας υπονομεύουν την διαγενειακή αλληλεγγύη και γενικά το κοινωνικό μας πρότυπο. Αυτό λοιπόν αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα κράτη-μέλη, οι διακρίσεις λόγω φύλου και ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη όπου είναι μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ε, θέλουμε μία βάση για καλή οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ε, θα ήταν λοιπόν χρήσιμο αυτά τα θέματα να δικατοπτρίζονται καλύτερα στις κατευθυντήρες γραμμές. Έχουμε τον ε, πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, καθώς και γενικά η συμμεταχείριση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τούμ, δεν βλέπω να είναι κανείς παρόν από την ΓΚΟΕ. Λάουρα, Ατζέα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Τζανόκα για την εργασία της. Εδώ και καιρό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό ε, έγγραφο και θέμα τις δύο προηγούμενες ε, φορές, τα δύο προηγούμενα χρόνια, ήμουν εισηγήτρια για αυτό το, για αυτό το σημαντικό έγγραφο. Και σημείωσα ότι παρά την μεγάλη δέσμευση, την γενική στράτευση στην Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποδυναμώθηκε η θέση, γιατί συχνά το Συμβούλιο αποφασίζει να αγνοήσει την εργασία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλά και αγνοεί στην ουσία και την ε, ε, ψηφοφορία και την βούληση που εκφράζεται μέσω της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Αναλύουμε λοιπόν ξανά το θέμα αυτό και ευελπιστώ η συνάδελφος ε, Τζανόκα να μπορέσει να ασκήσει όσο γίνεται μεγαλύτερη πίεση στο Συμβούλιο και την Κομισιόν έτσι ώστε οι ενδείξεις που υποβάλλουμε εμείς ως Κοινοβούλιο να ληφθούν υπόψη σε μεγάλο βαθμό. Είναι πολύ ε, ουσιαστικό ε, εμείς να έχουμε ένα κείμενο όσο γίνεται πιο ε, δυνατό έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αποδυνάμωσης του από την Κομισιόν ή από το Συμβούλιο. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι η Τατιάνα έλαβε υπόψη της και κάνει αναφορά στον κοινωνικό πυλώνα που βέβαια θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά με συγκεκριμένα μέτρα και και λόγω της ε, κοινωνικής ε, ε, επικινδυνότητας ας πούμε της ειδική κατάστασης που ζει η Ευρώπη αυτή την περίοδο. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τα μεγάλα λόγια και τα παχιά λόγια αλλά ε, συγκεκριμένες δράσεις το Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε το κείμενό μου για την ε, πολιτική υπέρ ε, της, ε, του ελάχιστου εισοδήματος και νομίζω ότι μαζί με το κείμενο της Αττιάνας αποτελούν πολύ σημαντικά κείμενα για αποτελεσματικές κοινωνικές πολιτικές. Θα πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσουμε σε συμπεριληπτικά και ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και βεβαίως ε, να βοηθήσουμε την διαβίου κατάρτιση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και τις υφιστάμενες ανάγκες αλλά και τις μελλοντικές ε, ανάγκες ε, της αγοράς εργασίας. Η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις συγκεκριμένες και ουσιαστικές κυρίως στους τομείς που αποτελούν ομοχλό της οικονομίας, την κοινωνική, κοινωνική συγγνώμη, κυκλική οικονομία, την πράσινη πράσινη οικονομία κτλ. Ε, οποτεδήποτε γίνονται αυτές οι επενδύσεις ε, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι αυτός ε, ο περιορισμός του 3%. Το θέμα της εργασίας βεβαίως ε, είναι πολύ σημαντικό γιατί η έλλειψη εναρμονισμένων φορολογικών πολιτικών και η φορολογική πίεση δημιουργεί πρόβλημα στην Ευρώπη και μεταφέρει, την μετατοπίζει την φορολόγηση σε άλλους τομείς ε, η Ευρώπη θα πρέπει οπωσδήποτε να οδηγηθεί ε, την, ε, στη χρήση ενεργειών που δεν παράγουν διοξίδιο του άνθρακα. Θα πρέπει να βοηθήσουν την ενεργειακή μετάβαση. Χρειαζόμαστε γενικά υπηρεσίες προσβάσιμες αλλά και προσιτές. Στέγαση και προστασία των ηλικιωμένων. Θέλουμε όλοι να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ε, υγείας, υγιεινής, αποχέτευσης, εκπαίδευσης, εργασίας. Ε, το 2018 στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να σκεφτούμε ότι αυτά τα βασικά δικαιώματα παραβιάζονται. Για τις στατιστικές ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί ε, δεν θεωρώ ότι ε, με την επιμήκυνση της εργασιακής ζωής θα λύσουμε οποιαδήποτε προβλήματα. Εάν οι νέοι δεν καταφέρουν να μπουν, να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει, να διατηρηθεί το συνταξιοδοτικό σύστημα. Υπενθυμίζω επίσης ε, ότι είναι ε, σημαντικό η συνταξιοδότηση κυρίως ε, για τα βαρέα και ανθυγιεινά ε, ε, επαγγέλματα η συνταξιοδότηση να γίνεται μάλιστα πιο νωρίς. Δεν είναι δυνατόν να μην συνταξιοδοτούνται νωρίτερα κάποιες κατηγορίες βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Οπωσδήποτε θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτό που εγώ ονομάζω διαγενειακή σκητάλη. Θα πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν και μια ευελιξία κατά αυτήν την έννοια Ρουμανία έτσι ώστε να επιτρέψουμε στους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας. Τέλος, θα πρέπει ε, να βοηθήσουμε, την, ε, ε, να βοηθήσουμε τους νέους, να διευκολύνουμε το turnover στην εργασία και να βοηθήσουμε και τους πιο ηλικιωμένους να εγκαταλείψουν την εργασιακή ζωή. Να σκεφτούμε τους ηλικιωμένους, να σκεφτούμε τους εργαζόμενους, των οποίων τα χρόνια περνάνε και κάνουν αυτά τα λεγόμενα βαρέα και ανθικά ανθυγιεινά επαγγέλματα ε, και ε, θα πρέπει να, έχουμε, να έχουν αυτή τη δυνατότητα να πάρουν σύνταξη πιο νωρίς. Αυτά ε, θα είναι τα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν στοιχεία για τα οποία εγώ θα υποβάλω τροπολογίες έτσι ώστε να γίνει ένα κείμενο δυνατό για να υποχρεώσουμε, να πιέσουμε το Συμβούλιο να λάβει υπόψη το κείμενο. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου του ΙΕΝΕΦ, ο κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Όσον αφορά αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόληση των κρατών μελών που διατυπώνονται κάθε χρόνο, ε, δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπα και πριν από μερικέ εβδομάδες. Τέλο πάντων, χοντρικά είχα πει ότι πρόκειται για ένα κατάλογο ευσεβών πόθων. Φυσικά και είμαστε υπέρ επί της ουσίας, γιατί όλοι θέλουν την πλήρη απασχόληση. Αλλά το χειρότερο είναι ότι υπενθύμησε, το υπενθύμησε και η Λόρα Αζέα, πρόκειται για ευσεβείς πόθους που όμως δεν λαμβάνονται τελικά υπόψη ούτε από την Επιτροπή ούτε από το Συμβούλιο. Οπότε, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ σήμερα το πρωί τόσες ώρες εργασίας κάθε χρόνο για αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Τα είπα και πριν από μερικές εβδομάδες. Τώρα κύριε Συγκίτρια, παρά τις κάποιες καλές σας προτάσεις, για τις οποίες σας ευχαριστώ, βλέπουμε διάφορες τροπολογίες που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Για παράδειγμα, να συμπεριληφθεί ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τροπολογίες 5 και 11. Δεν βλέπω τι δουλειά έχουν εδώ. Όπως και ένταξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Και επίσης, εδώ λέμε τι προτιμάμε. Προτιμάω την ανιψιά μου από την ε, ξαδέρφη μου ή από τη γειτόνισσα που δεν ξέρω εγώ τι. Για μένα η προτίμησή μου πρέπει να δοθεί στους Γάλλους εργαζόμενους. Έπειτα υπάρχει και τροπολογία για μέτρα υπέρ των ε, προσφύγων και των υποεκπροσωπούμενων ε, κατηγοριών. Αυτή είναι δικιά σας επιλογή. Εμείς έχουμε 6 εκατομμύρια ανέργους στη Γαλλία και 9 εκατομμύρια που βρίσκονται κάτω από το όριο της στόχιας. Στη Γαλλία, ε, και τα έχουμε τα ίδια και στην Ιταλία και στην Ισπανία, ακόμα και στη Γερμανία. Μας λένε για τη Γερμανία κάθε τόσο, ναι, αλλά αμοιβέ στη Γερμανία είναι αστείε. Οπότε, αν πρόκειται για προτίμηση, εμεί έχουμε την εθνική προτίμηση, κυρία Συγκίτρια. Οπότε και εμεί θα υποβάλουμε τροπολογίε προ αυτή την κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Ήμουνα σύντομο, ε. Πρόεδρο, ναι, πράγματι, πολύ σύντομο. Πράγματι. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα και άλλος ο κύριος Μαρτάν όμως έχει ζητήσει το λόγο. Οπότε εσεί τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, Εντουάρι είναι το μικρό μου, οπότε... Λοιπόν, έχω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις για τις κατευθυντήριε γραμμές. Πώς θα έπρεπε να είναι αυτές. Θα έπρεπε να τονίσουμε και το θέμα της μείωσης του χρόνου εργασίας. Εγώ χαίρομαι για την συμφωνία της Αγγε Μετάλ στη Γερμανία που λέει ότι από... μπορούμε να περάσουμε κάτω από κάποιες προϋποθέσεις τις 28 ώρες τη βδομάδα. Πιστεύω και εγώ ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Δεν μιλάμε για την ψηφιοποίηση, ρομποτική κτλ. Οπότε πρέπει να δούμε και πώς θα γίνει η κατανομή του πλούτου. Και όταν μιλάω για τη μείωση του χρόνου εργασίας, εδώ παίζει και ε, το θέμα της ηλικής ταξιδότησης. Γιατί συμφωνώ με την Ιταλίδα συνάδελφο, δεν μπορεί να λέμε θέλουμε την πλήρη απασχόληση και απ' την άλλη να κρατάμε τον κόσμο στη δουλειά όσο γίνεται περισσότερο. Και έρχομαι τώρα στους νέους και την κατάρτισή τους. Ε, κάποιες χώρες το έχουν εγκαταλείψει. Ε, στη χώρα μου πριν από κάποια χρόνια ε, είχαμε ουσιαστικά κλείσει την επαγγελματική εκπαίδευση και είχαμε μιζάρει σε μακροχρόνιες σπουδές, ότι όσο πιο πολύ σπουδάζει κανείς τόσο το καλύτερο, αντί να εκπαιδεύσουμε τους νέους στην επαγγελματική κατάρτιση. Γιατί σε πολλές χώρες και στη Γαλλία και όχι μόνο, δεν υπάρχει αρκετή κατάρτιση για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της αγοράς. Η διαβίου μάθηση τώρα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τα είπαμε λίγο χτες στη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Τάισεν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το δικαίωμα στην κατάρτιση διαβίου. Και τώρα επειδή τα πράγματα δεν γίνονται μηχανικά, μπορεί να καταργήσουμε θέσεις απασχόλησης σε κάποιο σημείο και να υπάρχει ζήτηση κάπου αλλού ναι, αλλά ανάμεσα στα δύο μπορεί να μεσολαβούν εκατοντάδε χιλιόμετρα. Άρα πρέπει να υπάρχει και βοήθεια στην κινητικότητα, γιατί μπορεί κάποιο να θέλει να φύγει από την περιοχή που ζει και να πάει κάπου αλλού αν έχει εκεί δουλειά, αλλά χρειάζεται κάποια βοήθεια για αυτή την κινητικότητα. Πρέπει να το προβλέψουμε και αυτό, συνεπώς. Έτσι θα βοηθήσουμε να υπάρξει αυτή η αντιστοιχία. Αυτά είχα να πω επιπλέον από τόσα προτάθηκαν, αλλά σίγουρα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Εντουάρ Μαρτά. Τώρα, δεν βλέπω κανέναν άλλον να θέλει το λόγο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να σχολιάσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ, πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι κατευθυντήριες γραμμές είναι πάρα πολύ σημαντικές από θεσμικής πλευράς, διότι παρέχουν τη νομική βάση αποτελούν δηλαδή μια νομική βάση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το ε, Συμβούλιο κάθε χρόνο. Ε, αποτελούν όμως και τη βάση για τις συστάσεις αναχώρα όσον αφορά την απασχόληση. Φέτος ε, με τις προτάσεις αυτές προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε πλήρως την ε, διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που είναι κάτι που έχει γίνει όχι μόνο από τα κράτη-μέλη αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συχνά λοιπόν έχουμε παραθέσει ακριβώς το κείμενο των αρχών του πυλώνα. Εάν αυτό δεν ήταν δυνατόν προσπαθήσαμε να παραμείνουμε όσο γίνεται πιο κοντά στο κείμενο αυτό. Προσπαθήσαμε λοιπόν όπου είναι δυνατόν να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία. Η λογική αυτή φαίνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεώρησα σημαντικό να το επισημάνω. Δεν ε, θέλω αυτή τη στιγμή να σχολιάσω εις βάθος ε, το σχέδιο έκθεσης. Απλά ήθελα να επισημάνω ποια είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε, δηλαδή ότι ακολουθούμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα ε, ε, κοινωνικών δικαιωμάτων ε, και ότι αυτός χρησιμοποιείται και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι σημαντικό ότι τον πυλόν αυτό θα πρέπει να τον υποστήριξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω την εισηγήτρια, αν θέλει να σχολιάσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς τους εσκιώδεις εισηγητές. Συμφωνώ με τις περισσότερες παρατηρήσεις. Ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις της Λάουρα. Έχουμε αλλάξει θέσεις. Ήταν εκείνη η εισηγήτρια και ο Σκιώδης, ενώ τώρα έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Πολύ με Πολύ αισιοδοξία μου προκαλούν και τα ε, ε, λόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα λάβετε υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου στις νέες κατευθύντες γραμμές. Ο κύριος Ντομινίκ Μαρτέ. Ε, ναι, έχουμε σύγχυση ως προς το επώνυμο Μαρτέ αναφέρθηκε στην ε, τροπολογία 31 για την ε, κατευθυντήρια γραμμή 8 ε, και τις μη διακρίσεις. Φυσικά έχουμε διαφορετική πολιτική θέση, είναι γνωστή η θέση μας. Και ήμουν εισηγήτρια το 2006 του Κοινοβουλίου σχετικά με την στρατηγική μας θέση για τις μη διακρίσεις και ήταν και η εποχή το 2007 που είδαμε τα προβλήματα στην Γαλλία όπου επισήμως ε, δεν γίνονται διακρίσεις, αλλά είδαμε διακρίσεις εις βάρος μιας ομάδας του πληθυσμού. Ελπίζω λοιπόν οι περισσότερες πολιτικές ομάδες να στηρίξουν την πρόταση αυτή μετανάστες, ε, ε, εθνοτικές μειονότητες και άλλες ε, ομάδες μειονοτήτων να μην γίνονται θύματα διακρίσεων. Αποφάσισα να εγκαταλείψω τη θέση μου πριν την λήξη της θητείας, ε, διότι θα είμαι υποψήφια σε εκλογές. Η έκθεση αυτή θα... την έκθεση αυτή θα αναλάβει ο συναδελφός μου που είναι και έμπειρος ε, και σας εύχομαι καλή συνέχεια των εργασιών. Πρόεδρος, είναι η τελευταία σας ε, συνεδρίαση στην Επιτροπή Απασχόλησης. Θα είμαι εδώ την επόμενη εβδομάδα. Ωραία λέει Πρόεδρος, ε, θα αποχαιρετιστούμε τότε στην επόμενη συνεδρίαση. Κρίμα που δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε τις εργασίες πάνω στην έκθεση αυτή. Αλλά βέβαια καταλαβαίνω την ε, επιλογή σας. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 28 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Όποιο θέλει λοιπόν να υποβάλει τροπολογίε α γνωρίζει την προθεσμία. Εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στη συνεδρίαση τη ΕΜΠΛ 21 ε, και 22 Μαρτίου. Θα ψηφίσουμε την έκθεση 25-26 Απριλίου η έκθεση φυσικά θα παραμείνει, θα διατηρήσει το πνεύμα σας παρότι δεν θα είστε πια παρούσα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι το 17 έχει αναβληθεί. διότι οι άνθρωποι που ήταν να μας παρουσιάσουν την έκθεση δεν κατάφεραν ε, να ε, μεταβούν λόγω ε, απεργίας Ω προερχόμενη από συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει να επικροτήσω την απεργία φυσικά, αλλά ναι. Η επόμενη συνεδρίασή μα θα πραγματοποιηθεί 26 και 27 Φεβρουαρίου. Εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που θέλουμε να θίξουμε, λίγη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ.